Ο κύριος Μπάρι Μάτλενερ μου ε, γνωστοποίησε την παρέτησή του από μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 20 Σεπτεμβρίου 2012. Το Κοινοβούλιο διαπιστώνει ε, τη χειρία της θέσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού. Οι αρμόδιες αρχές ε, των κάτω χωρών με ενημέρωσαν ότι από την 3η Οκτωβρίου 2012 ο κύριος Μάτλενερ ε, αντικαθίσταται από την κυρία Πατρίσια Βάντερ Κάμεν. Καλώς ορίζω τη νέα συνάδελφο και σημίζω ότι η κυρία Βάντερ Κάμεν σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού απολαμβάνει τη δυνατότητα να συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα στη συνεδριάση του Κοινοβουλίου και των Επιτροπών σε περίπτωση ε, και με την προϋπόθεση ε, ότι ε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ασυμβίβαστου με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτού και εφόσον ε, δεν έχουν ελεγχθεί ακόμα ε, τα διάφορα δικαιολογητικά.